Liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση, που μπορεί να είναι από τις τελευταίες συνεδριάσεις, αλλά και μία από τις σημαντικότερες, διότι σήμερα θα συζητήσουμε την τελική έκθεση της Περβάνς που είναι η αρμόδια εισηγήτριά μας και μάλιστα εκτενώς θα τη συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Πριν δώσω το λόγο στην Περβάνς Μπερές για να μας παρουσιάσει τα βασικά σημεία της έκθεσής της θα ήθελα, μου επιτρέπετε, να σας κάνω δύο ανακοινώσεις στο σημείο 2 της ημέρησια διάταξης μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά για την αντιπροσωπεία μας ε, που πριν από μια εβδομάδα Ακριβώ Δευτέρα και Τρίτη πήγε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα της Επιτροπής μας στο τελευταίο δελτίο της γραμματείας που είναι τώρα επί του πιεστηρίου θα διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη αυτή της αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, αποστολή όσο και παραγωγική. Είχαμε επαφές με προσώπους κυβέρνησης, των τραπεζών, ομίλων, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επόμενη μέρα και με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά εκτός αυτού σχεδόν όλο το πρωί, την Τρίτη συγκεκριμένα, συναντήσαμε και συζητήσαμε με συναδέλφους από τη Βουλή των Ελλήνων, εκπροσώπους τριών επιτροπών οικονομικών, ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής και χρηματοπιστωτικών υποθέσεων. Ήταν πολύ ε, καλή η ανταλλαγή απόψεων και έδειξε το εξής. Και λυπάμαι γι' αυτό προσωπικά, ότι δηλαδή οι Έλληνες πολιτικοί εκπρόσωποι είναι βαθύτατα διχασμένοι για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Και αυτό που τους ευχήθηκα εγώ στην αρχή της τοποθέτησής μου ήταν να ξεπεράσουν όσο γίνεται να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές τους και εμπολείς ιδεολογικές τους διαφορές για να κατανοήσουν ότι το θέμα είναι εθνικό και από κοινού θα πρέπει να κάνουν ό,τι χρειάζεται, όπως έκαναν οι Σουηδοί τη δεκαετία του 90. Αυτό δυστυχώς φαίνεται αδύνατο στην Ελλάδα. Και στην Πορτογαλία από ό,τι είδαμε πρόσφατα είναι αδύνατο. Και φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των χρηματαγορών. Να ξανακερδίσουν δηλαδή την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών το βλέπω δύσκολο. Ακόμα και αν έχει βοήθεια αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και δεχομένω σε λίγε εβδομάδε και η Πορτογαλία να μπει στο μηχανισμό στήριξη, παρόλα αυτά φοβάμαι ότι η κρίση αυτή δεν έχει ε, διασκεδαστεί και ξεπεραστεί. Αυτά για την Αθήνα, τα υπόλοιπα παρακαλώ να τα διαβάσετε. Ε, συναντήσαμε και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ε, συνάντηση αυτή. Κατά τα άλλα, πρέπει να σας πω ότι τον Οκτώβριο είχαμε την διάμεση έκθεση, σήμερα έχουμε την τελική έκθεση και θα συζητήσουμε. Σκεφτήκαμε και είπαμε ότι θα ήταν μεγάλο κρίμα, μέχρι και ανευθυνότητα, Εάν όλα αυτά τα έγγραφα, ε, αναλύσεις, μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο, ε, αυτόν τον 1,5 χρόνο ζωής της Επιτροπής μας, να το αφήσουμε να χαθούν όλα αυτά τα πολύτιμα στοιχεία σε συρτάρια. Και η κοινή γνώμη να έχει μόνο πρόσβαση στην ενδιάμεση έκθεσή μας και σε τούτη εδώ την τελική. Γι' αυτό ε, συνεννοηθήκαμε εσωτερικά με την εισηγήτρια και με πολλούς άλλους συναδέλφους και τη γραμματεία βεβαίως κυρίως και αποφασίσαμε μετά το πέρας των εργασιών να κυκλοφορήσει ένα συμπίλημα που θα περιλαμβάνει ε, όλα τα έγγραφα τα θεματικά έγγραφα που είχαμε από την αρχή, τα πρακτικά ε, των αποστολών, των αντιπροσωπιών, πώληση και briefing papers, όλο αυτό το υλικό να το εκδώσουμε σε ένα ή δύο τόμους, να το τυπώσουμε για να έχουμε μια καθαρή βάση αναφοράς και να μπορεί κανείς να ανατρέχει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αν είναι ένα ή δύο τόμοι, ε, δεν θα είναι κάτι που θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, όσο συναρπαστικό και αν είναι για κάποιους, αλλά θα είναι μια καλή αναφορά για να μπορεί να τρέχει κανείς όταν το χρειάζεται. Και αυτά θα τα στείλουμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια και σε όλους εκείνους που θα ε, απευθυνθούσε μάλλον όλους όσοι μας ε, συμβούλευσαν, μας βοήθησαν στη δουλειά αυτή με στοιχεία και έγγραφα. Αυτά. Και έρχομαι τώρα στο σημείο 3 και θα δώσω το λόγο στην Περβάνος Περές να μας παρουσιάσει σύντομα παρακαλώ την έκθεσή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης, από ό,τι φαίνεται λίγα πράγματα έχουν επιληθεί και τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς κατευθύνσεις που κανένας σε αυτή την αίθουσα και ίσως και έξω από την αίθουσα είχε ποτέ φανταστεί πριν από τρία χρόνια. Και εμείς σήμερα φέρουμε μία ευθύνη ως προς αυτό που θα αποστείλουμε ως μήνυμα. Πριν έρθω στο, σχέδιο, στο τελικό σχέδιο της έκθεσής μου, Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μερικά σε αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς. Εγώ στην Αθήνα δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα διότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης ε, ε, μιλούσα στην ΔΟΕ σε μία συζήτηση που αφορούσε στις επιπτώσεις της Αραβικής Άνοιξης και της συνένεσης των Βρυξελών. Ε, και θα σταθώ σε αυτό που είπατε για την έλλειψη συνένεσης ε, στην Αθήνα και που σας εκπλήσει υπάρχει ένας προσανατολισμός στο Συμβούλιο και στις ε, προτάσεις ε, της Κομισιόν ένας προσανατολισμός που, προσανατολισμός που οδηγεί τις ε, χώρες σε μέτρα λιτότητας τα οποία δεν καταλήγουν σε γενική συμφωνία και το βλέπουμε παντού αυτό. Επίσης, χαίρομαι που μπορούμε να συντάξουμε τα άπαντα των εργασιών μας. Μπορούμε να έχουμε ίσως και τον λόγο του Ζακ Ντελόγ όταν απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια που ο λόγος ήταν στα αγγλικά βέβαια και αν θα πρέπει να δημοσιεύσουμε τα άπαντα των εργασιών μας Νομίζω ότι στα απαντά αυτών των εργασιών θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και ο λόγος του Ζαντελό. Τώρα επανέρχομαι στο κείμενο της έκθεσής μου. Αυτό το σχέδιο τελικής έκθεσης όλοι σας θα το καταλάβετε, είναι καρπός μίας διαφορετικής προβληματικής στις εργασίες μας. Εγώ χρησιμοποίησα όλο το υλικό και τις συνεισφορές των πολιτικών ομάδων και προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τις βασικότερες ανησυχίες οι οποίες ε, εγώ θεώρησα ότι μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση συνένεσης. Μερικές παρατηρήσεις τις έχουμε στην εισαγωγή της έκθεσής μου. Για κάποια εμπόδια τα οποία το ρίσαμε μαζί. Θα έπρεπε να δούμε την εντολή μας στο δεύτερο τμήμα των εργασιών μας και η οποία εντολή συνίστατο στο να διαπιστώσουμε πώς γινόταν αντιληπτές οι προτάσεις μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια και δεύτερον πώς οι προτάσεις που επεξεργαστήκαμε αρχικά θα έπρεπε να επεξεργαστούν για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Δεν σας προτείνω να ανοίξουμε τα σημεία εκείνα τα οποία ήταν συνενετικά στην πρώτη έκθεση. Και δεν προτείνω να ανοίξουμε αυτά τα οποία οι συντονιστές είχαν ορίσει ως μέτρα που θα έπρεπε να αναλυθούν για την έξω από κρίση. Αυτά όμως ήταν μέτρα τα οποία ήδη ψηφίστηκαν στο Κοινοβούλιο το Μάρτιο για την ε, χρηματοπιστωτική καινοτομία. Δεν θα ξανανοίξουμε λοιπόν αυτά τα κεφάλαια. Επίσης έχουμε και άλλες νομοθετικές εργασίες ε, στα Σκαριά, εδώ στην, στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, στην Επιτροπή Ενέργειας. Στα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Και όσον αφορά και στις δημοσιονομικές προπτικές υπάρχει μια ειδική επιτροπή που εργάζεται γι' αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε παράλληλα. Για την ουσία της έκθεσης. Αν δούμε ποιο ήταν το βασικό μήνυμα γύρω από το οποίο υπήρχε συνένεση και ψηφίστηκε σε μεγάλη πλειοψηφία στις 20 Οκτωβρίου στο Κοινοβούλιο. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Και αυτή την εμβάθυνση πρέπει να την κάνουμε σε δύο επίπεδα. Παγκόσμια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της δεύτερης έκθεσης. Υπάρχουν θέματα για τα οποία αναγνωρίζω ότι αντιμετώπισα δισταγμούς και στη συζήτηση στην ομάδα εργασίας με τους ε, συναδέλφους ε, τι ήταν η συνένεση, διότι εμείς λέμε ναι χρειάζεται μια μεγαλύτερη παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά συμφωνούσαμε, αλλά τι κρυβόταν πίσω από όλα αυτά. Υπήρχαν δυσκολίες γιατί δεν είχαμε μεν και δε τις ιδέες ξεκάθαρες. Εγώ πιστεύω, βασιζόμενοι πάντα στην πρώτη έκθεση, ότι το βασικό μήνυμα θα μπορούσε να έχει ως εξής. Η κρίση προέρχεται από τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Άρα κατά συνέπεια πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Και φυσικά δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε μια παγκόσμια λύση που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες των μεν και των δε. Τώρα για την εφαρμογή αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τρία χρόνια μετά από την κρίση, οι μηχανισμοί παρακολούθησης των χρηματοπιστωτικών αγορών που συστήσαμε δεν μας επιτρέπουν να πετύχουμε την καλύτερη, το optimum στη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Και αυτό πρέπει να το, ε, να το καταλάβουμε. Και αυτό έχει άμεση επίπτωση στο θέμα του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Αλλά αυτό όμως τίθεται πάντα μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο που εγώ διαπίστωσα. Και όσον αφορά τώρα στις προκλήσεις του διεθνούς νομισματικού συστήματος, για τους Ευρωπαίους είτε είναι μέσα ή έξω από τη ζώνη ευρώ. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο θέμα των διαφορών ανταγωνιστικότητας. Και στο όνομα αυτών των διαφορών ζητάμε από τους διάφορους λαούς που υποφέρουν από αυτήν τη διαφορά ανταγωνιστικότητας να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες που μπορούμε να τις ονομάσουμε πολιτικές λιτότητας. Βλέπουμε επίσης κερδοσκοπικές κινήσεις επί των νομισμάτων και αυτές οι κερδοσκοπικές κινήσεις σβήνουν, διαγράφουν μια για πάντα όλες τις προσπάθειες. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να ασχοληθεί με και με το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Για το τέταρτο τώρα κεφάλαιο που έχει να κάνει με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναρωτιέμαι μερικά πράγματα. Και πολλές από αυτές τις ερωτήσεις κατάλαβα ότι μπορούμε να τις συμμεριστούμε όλοι μας είναι το θέμα των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των επενδύσεων για το μέλλον. Ε, μπορούμε εμεί επιτυχώς να φανταστούμε την εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 αν δεν συζητήσουμε το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εγώ δεν ικανοποιούμε με τη λύση που θα έλεγε ότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον χρήμα. Οπότε οι μελλοντικέ, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα βασιστούν στις μαζικές ροές ρευστού από την Κίνα ή από αλλού. Εντάξει, μπορεί να έρθουν αυτά τα κεφάλαια και να είναι καλόδεκτα. Αλλά δεν είναι αυτή η ευρωπαϊκή απάντηση που πρέπει να δοθεί για τη ροή των κεφαλαίων. Και αυτό λέει πολλά για τη στρατηγική που θέλουμε να εφαρμόσουμε για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, πιστεύω ότι και σε μία διακύμανση των ενιών της πρώτης έκθεσης θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα της εκπαίδευσης. Ε, όταν μιλάμε για εκπαίδευση δεν είναι η χρηματοδότηση Twitter, του Γαλιλαίου, ε, των τρένων υψηλής ταχύτητας. Όχι, είναι κάτι το λιγότερο ορατό, κάτι το υπόγειο. Αλλά από στρατηγικής πλευράς είναι πολύ πιο σημαντικό. Εγώ το λέω ειλικρινά. Δεν το γράφω έτσι στην έκθεση, αλλά σας το λέω για να τα έχουμε ξεκάθαρα τα πράγματα μεταξύ μας. Όταν εγώ βλέπω τα προγράμματα λιτότητας, ανησυχώ όταν ζητάνε δηλαδή από τις χώρες να συνεχίζουν τη στρατηγική για το 2020 και από την άλλη να βλέπω τους προϋπολογισμούς όπου λαμβάνονται ή λαμβάνονται υπόψη η χρηματοδότηση μέσω κεφαλοποίησης και δεν αναφέρεται τίποτα για τη χρηματοδότηση στην εκπαίδευση. Το βασικό μήνυμα λοιπόν που θεωρήσαμε ήδη από την πρώτη έκθεση ήταν το εξής το Κοινοβούλιο συμφώνησε να στην πρώτη έκθεση αλλά όπως είπε και ο Ζακ Ντελόρ στο λόγο του χωρίς ολοκληρωμένη συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και άμα δεν συμβεί, άμα δεν έρθει αυτό, τότε χρειάζεται η ενισχυμένη συνεργασία. Εγώ είμαι κατά της ενισχυμένης συνεργασίας, είναι κατά της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Αυτοί που σήμερα όμως είναι μέλη της ζώνης ευρώ έχουν μια ειδική ευθύνη, ιδιαίτερη ευθύνη και για τους ίδιους αλλά και για την Ευρώπη. Και το να παίρνει κανείς ο ε, ανάλογα με το αν είναι στη ζώνη ευρώ ή όχι, δεν μπορεί να αποτελέσει την προπτική της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Διότι και εμείς παγιδευόμαστε, αλλά και οι λαοί που επέδειξαν εμπιστοσύνη για το ενιαίο νόμισμα. Εγώ ξέρω ότι με 63 παραγράφους το κείμενό μου είναι ένα πυκνό κείμενο. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο να στείλουμε ένα σύντομο μήνυμα σαφές και να επιδείξουμε ευθύνη και ο αριθμός των τροπολογιών να είναι σε λογικά πλαίσια. Εγώ υπολόγισα γύρω στα 300 για να μπορέσω να τα εντάξω στην έκθεσή μου. Και να μπορέσουμε όλοι λοιπόν να επιδείξουμε ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Περβάνσου για την εισαγωγή αυτή και την παρουσίαση της έκθεσή σου. Ευτυχώς αυτή τη φορά είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην χρειάζεται να συζητήσουμε το σκελετό της έκθεσης. Συμφώνησαν οι συντονιστές για αυτά τα πέντε κεντρικά σημεία. Γι' αυτό και η δομή και η διάρθρωση. Και όπως είπες και στο τέλος, να έχουμε μια σύντομη σχετικά έκθεση με ε, σαφέστατο μήνυμα και ήδη νομίζω αυτά έχουν οριστεί εκ των προτέρων. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Να δώσω το λόγο σε εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, καταρχάς και μετά στα μέλη της Επιτροπής μας. Με τη σειρά λοιπόν, Φρανκέρ, Κοφεράτη, Όλε Σμιτ, Πασκάλ Καλφίν και ο Νίκος Οχουντής, εκπρόσωποι των συντονιστών και των πολιτικών ομάδων και μετά θα ανοίξει συζήτηση για Το τον είπα δεύτερο το κοφεράτη. Μην ανησυχεί περβάς. Ε, ε, euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζοντας θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς την εισηγήτρια. Ενσωμάτωσε, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, όλα τα ουσιαστικά στοιχεία των προτάσεών μας τη στιγμή που τις υποβάλαμε. Βέβαια, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι τρόπον την Α, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε ένα-δύο χρόνια τις εργασίες μας, διότι ακόμη δεν φτάσαμε σε ένα σημείο όπου να μπορούμε να πούμε ιδού η λύση για την έξοδο από την κρίση. Έχω την εντύπωση, ξαναλέω, ότι θα, μπορούσε, να, θα μπορούσαμε να χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτά που είχαμε προβλέψει προεξαμήνου ή δωδεκαμήνου ε, και η αποστολή που έγινε στην Ελλάδα επιβεβαίωσε αυτό μου το φόβο, αυτή την εντύπωση μάλλον, διότι διαπιστώνουμε ότι ανάλογα με το βάθος της ύφεση στο οποίο έχει βυθιστεί ένα κράτος ε, έχοντας χάσει τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών, μάλλον των δημοσιονομικών παραγόντων του, ε, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να επανέλθει μια χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει με τις πρόορες εκλογές επίσης στην Πορτογαλία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και πολλά πράγματα αυτό. Αλλά βλέπετε τι έγινε με τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια στην Ισπανία. Κανείς δεν ξέρει τελικά τι έγινε με τις ληξιπρόθεσμες αφιλές. Θέλουμε να αποφύγουμε ένα νέο μαζικό κύμα που δύσκολα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε με δημοκρατικό τρόπο, δηλαδή το κύμα αντίσταση ω προ την πυρηνική ενέργεια δεδομένου του ατυχήματο που έγινε. Ναι, μεν πολύ μακριά από την Ευρώπη, αλλά το οποίο μα απασχολεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε προχωρήσει και πολύ τον τελευταίο χρόνο για να συνοψίσω τη θέση μου. Ε, συγκροτούμε διάφορους μηχανισμούς για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε γιατί τη χαρακτηρίζουμε οικονομική αυτή τη διακυβέρνηση, ούτε σε τι έγκυται αυτή η διακυβέρνηση. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε καταλήξει πάντως ε, σε συμπεράσματα που μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Ε, από πλευράς χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής εποπτείας αναρωτιέμαι επίση πώς ακόμη θα μας χρειαστούν αν τελικά η έκβαση των πραγμάτων στην Ελλάδα είναι χειρότερη από τα αναμενόμενα. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο και πληγεί ο τραπεζικός τομέας ε, στην Ελλάδα, θα μπορούσε να εκραγεί εκ των έσω ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η πρόκληση και νέα, διότι δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά όπως θα λέγανε και οι Ιαπωνές δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει όλα. Για το ίδιο το σχέδιο έκθεσης θα έλεγα ότι είναι καλό το μέγεθος. Τώρα για τη δομή νομίζω έχουμε συμφωνήσει όλοι, έχουμε συνενέσει για τη δομή. Είναι ορθή και πιστεύω ότι θα πρέπει επ' αυτού να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Μέσα στο σχέδιο έκθεσης επιδοκιμάζουμε τις ε, προτάσεις εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διότι διαπιστώνουμε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς σε ποιον άλλο τομέα παραδείγματο χάρη. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποτίθεται ότι πρέπει να ασχολείται με τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ, τελικά τι κάνουμε, λέμε α είναι χαλεπή η καιρή, δεν θα μα στηρίξει ούτως ή άλλως το Συμβούλιο. Οπότε λέει η αλλω είμαι συνετή. Ε, εξ αρχής, ε, συγκρατημένη εξ αρχής. Είναι πλημελέστατη αυτή η επιτροπη θα ειμαι συνετη εξ αρχή, συγκρατημενη εξ αρχη ειναι πλημελεστατη αυτη η σταση κυριω για το Κοινοβούλιο, διότι δεν είναι ο δικό μα ο ρόλος να είμαστε προσεκτικοί, συνετοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε φιλόδοξοι, γιατί άλλοι δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι. Οπότε, μέσα από τις φιλοδοξίες μας ενδεχομένως να καταφέρουμε να επηρεάσουμε την, το νου των πραγμάτων ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, ε, σε αυτό το στάδιο, Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι ε, η δική μου η πολιτική ομάδα δεν θα έχει σοβαρά προβλήματα. Θα περιοριστούμε ε, στις τροπολογίες μας ε, δεν θα υποβάλουμε υπερβολικά πολλέ. τουλάχιστον ελπίζουμε η συγγήτρια να θεωρήσει ότι είναι διαχειρίσιμος ο αριθμός των τροπολογιών που θα υποβάλουμε. Εγώ αναλαμβάνω δέσμευση προσωπική να μην κατευθυνθούμε προς τις 500 τροπολογίες. Ε, καμιά δωδεκαριά, ε, κάποιες ντουζίνες τροπολογιών νομίζω μπορούμε να τις ε, διαχειρίσουμε. Θα παραμείνουν υπό έλεγχο και μπορούμε να εργαστούμε έτσι νομίζω. Και στις 12-13 Απριλίου, πότε είναι που θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή μας, θα δούμε σε ποια λύση θα έχουν καταλήξει οι πολιτικές ομάδες. για αυτό το θέμα. Αν κατάλαβα καλά, ε, τα μέτρα που έχουν αποφασίσει άλλες εθνοσυνελεύσεις για την έξοδο από την κρίση, θεωρώ ότι οι δικές μας προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι πληρέστερες διεξοδικότερες σε σχέση με αυτά που έκαναν συνάδελφοι από άλλε εθνοσυνελεύσει, βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη ότι είχαν και εντελώ διαφορετική εντολή από εμά. Ευχαριστούμε. Φράνκο Σέρς Κομφεράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να δικαιολογήσουν ε, την απουσία πολλών σοσιαλιστών συναδέλφων γιατί συνεδριάζει η ομάδα αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα και υπάρχει μία αντικειμενική δυσκολία, υπάρχει μία συμβατότητα δηλαδή χρόνου. Και θα κοιτάξουμε να τους αντικαταστήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και το λέω αυτό γιατί η ομάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ε, τελική, για την ολοκλήρωση δηλαδή της συζήτησης της έκθεσης ε, της Περβάνσου. Η απουσία έχει να κάνει δηλαδή με λόγους υποδομής ε, και όχι με, για λόγους ουσίας. Προσθέτω Προσθέτω έλεγα ό,τι θα κάνω, ό,τι περνάει από το χέρι μου για να περάσει η έκθεση της Περβάος και από τη σοσιαλιστική ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό τροπολογιών. Διότι με λίγες τροπολογίες μπορούμε να εμπλουτίσουμε κάτι το οποίο σημεριζόμαστε όλοι μας και θα πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε ένα μια υπερβολή προσθήκων που θα αποδυναμώσουν το κείμενο. Πρέπει να βοηθήσουμε την εισηγήτρια και γι' αυτό. Είναι απόλυτα αποδεκτή η πρόταση της Περβάνς. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε σε αυτή τη σύσταση με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πολύ σημαντική η μεθοδολογική, η μεθοδολογική διάσταση που εγκρίναμε. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ένα πιο συνθετικό κείμενο, πιο ελαφρύ και πιο εύχριστο στο μέλλον. και να μην ε, επανερχόμαστε σε θέματα τα οποία ήδη συζητήθηκαν στην Επιτροπή μας και ήδη έχουν περάσει από την Ολομέλεια. Και αυτή η επιλογή θα μας βοηθήσει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αντικειμενικές δυσκολίες που δεν εξαρτώνται από μας. Όπως έλεγε ο συνάδελφος Έγγελς, η κρίση δεν τέλειωσε. Τουναντίον, σε, σε επόμενες εβδομάδες μπορεί να έχουμε νέα προβλήματα ή αναπαραγωγή προβλημάτων σε χώρες που μέχρι τώρα ήταν προστατευμένες από την κρίση. Είδατε τι έγινε στην Πορτογαλία. Κανένας όμως δεν μπορεί να αποκλείσει απριορί ότι και άλλες χώρες θα μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι. Βέβαια τα μέτρα για, για να αντιμετωπιστεί η πορτογαλική κρίση είναι διαφορετικά από εκείνα που εγκρίθηκαν για την Ελλάδα ή την Ιταλία και αποτελούν τον καρπό ε, των εργασιών αυτής της Επιτροπής και των υποδείξεων που δώσαμε. Και αυτές οι υποδείξεις βοήθησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν με διαφορετικά μέσα και με μια διαφορετική αποτελεσματικότερη μέθοδο τις ε, δυσκολίες της Πορτογαλίας. με πείθει ιδιαίτερα το πλαίσιο που μας υπέδειξε η Πρέπει να βγούμε από την κρίση δίνοντας μια νέα όθηση στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, μοντέλο το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες με διάφορους ε, τρόπους και μορφές. Πρέπει να θεωρήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ως σημαντικότατο παράγοντα, όπως επίσης και την άσκηση προληπτικών πολιτικών. Αλλά η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι εγκυμένη μόνο από την ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα. Διότι αν δεν υπάρχει ανάπτυξη δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Στόχος μας είναι πάντα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Και αυτό το μοντέλο αποτελεί ταυτότητα για μας, για την Ευρώπη. Είναι το χαρακτηριστικό μας και πρέπει να δούμε και μακροπρόθεσμα. Βέβαια η τελική μας, ε, το τελικό μας διάβημα θα έχει ακόμα πολλές αβεβαιότητες και η Περβάος ανέφερε μία από τις προτεραιότητες ε, για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Οι δραματικές, ε, οι περιπέτειες στη Ιαπωνία, η κρίση στην Βόρεια Αφρική θα ξαναγράψουν όλο το κεφάλαιο για την ενέργεια, για την προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. Θα διαμορφώσουν νέες σχέσεις μεταξύ των χωρών που έχουν αυτές τις πρώτες ύλες και των χωρών που θα πρέπει να τις προμηθευτούν. Δηλαδή, το πώς θα αξιολογήσουμε στο μέλλον την πυρηνική ενέργεια, πώς θα ορίσουμε την προμήθεια από τις παραδοσιακές πηγές καυσίμων, ας πούμε το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, πώς θα οριστούν οι τιμές τους στο μέλλον. Θα υπάρξουν δηλαδή στοιχεία αλλαγών τα οποία θα χαρακτηρίσουν το μέλλον. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να κοιτάξουμε μακριά και να προτείνουμε ένα, μια νέα ιδέα μοντέλου ανταγωνιστικότητας διαφορετικό από αυτό που είχε προταθεί μέχρι σήμερα στο Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ιδιαίτερα πιστική την επιλογή στόχων. Τόσο δηλαδή που αυτοί οι στόχοι ήδη έχουν ουσία, έχουν όμως και μια συμβολική αξία. Το θέμα της εκπαίδευσης το σχολείο το οποίο οδηγεί σε διάφορα επίπεδα γνώσης. Η γνώση που οδηγεί στην κοινοτομία και στην έρευνα αντικειμενικά θα πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ενός μοντέλου ανταγωνιστικότητας βάσει του οποίου η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και έχει δίκιο η όταν λέει το να ζητήσουμε από έναν αρχηγό ε, κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση σε μία φάση κρίσης δεν είναι εύκολο. Μα ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο είναι πολύ σημαντικό γιατί οι μεγάλες στρατηγικές λύσεις βρίσκονται όταν έχουμε δυσκολίες, όταν βρισκόμαστε σε στενοπούς, όταν δεν έχουμε ε, την δυνατότητα. Και εμείς θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προσπάθεια των κρατών μελών. Και το είπαμε αυτό και στις συζητήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία ταυτότητας της ευρωπαϊκής κουλτούρας άσχετα από το ανήκειν σε οποιαδήποτε πολιτική οικογένεια. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα πρέπει να καταγραφούν στην τελική έκθεση σαφέστατα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αποδώσω τα εύσημα στην εισηγήτρια πρώτα απ' όλα. Παρότι δεν είμαστε στην ίδια πολιτική οικογένεια και ορισμένες φορές διαφωνούμε σε μεγάλο βαθμό, παρόλα αυτά έκανε πολύ καλή δουλειά και θέλω να το αναγνωρίσω. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και εμείς προσπαθήσαμε να σας δυσκολέψουμε το έργο σας έτσι περαιτέρω. Θέλω να πω κάτι για την ε, Ελλάδα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αποστολή αλλά και λίγο απογοητευτική. Εάν οι πολίτες, εάν οι άνθρωποι δεν επιθυμούν την αλλαγή, δεν μπορούμε ε, από τις Βρυξέλλες να την επιβάλλουμε, ούτε καν από το Βερολίνο. Ήταν λοιπόν μάλλον απογοητευτική η αποστολή. Δεν χρειάζεται τον να κηρύσουμε εδώ, αλλά αν επιθυμούμε μια Ευρώπη που θα ενεργεί από κοινού, η πολιτική του Κοινοβουλίου και η πολιτική των κρατών μελών πρέπει να δρουν με ιδιαίτερα υπεύθυνο τρόπο και διαβλέπω κάποιες τάσεις που διαψεύδουν αυτή τη θεωρία σήμερα. Είναι ανησυχητικό, τουλάχιστον για μένα. Νομίζω ότι από χώρα εκτός ε, ζώνης ευρώ έχουμε ένα συντονιστή μόνο εμένα Εντάξει, βέβαια η χώρα μου δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ε, ζώνη του ευρώ και άρα ίσως δεν ξέρετε πώς να τις όλες αυτές τις παρατηρήσεις που κάνω. Ε, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα εν τέλει, αλλά θέλω παρόλα αυτά να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, συμφωνήσαμε ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια κοινή πλέον προσέγγιση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η έκθεση με ακρίβεια τον αναφέρει, αλλά περιγράφει και ένα όραμα για το μέλλον. Ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης σήμερα είναι το εξής. Όταν εγώ πρώτον μπήκα στην πολιτική, είχα από τότε ένα φίλο και μου είπε ότι οι ηγέτες πρέπει να καθοδηγούν το λαό, να εκφράζετε τις επιθυμίες σας, αλλά δεν μπορείτε να κινήσετε τόσο γρήγορα που να εξαφανίσετε και να μην σας βλέπουν καν οι να μην σας βλέπουν οι πολίτες. Ενώ αυτό είναι το πρόβλημα του Κοινοβουλίου και θα πάρω ένα ε, παράδειγμα ε, συγκεκριμένο. Πέρσι, στον προϋπολογισμό, όλα τα κοινοβούλια, όλοι οι συνάδελφοι στην Ευρώπη ε, είχαν τα μέτρα της ε, λιτότητας. Εμείς όχι πάλι. Εμείς μεγαλώσαμε τα ποσά, τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Αυξήσαμε τον προπολογισμό. Καλές ήταν οι προθέσεις, δεν λέω, αλλά ήταν καταστροφικό το αποτέλεσμα και υπέθαλψε και τον ευρωσκεπτικισμό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού, ότι δεν είμαστε τόσο κοντά στους πολίτες όσο θα θέλαμε. Κάποιοι συνάδελφοι στις πρωτεύουσες είναι πολύ κοντύτερα στους πολίτες, πολύ εγκύτερα. Έχω κάποια σχολεία για αυτή την λίαν ομοσπονδιακή θεώρηση των πραγμάτων. Κάθε παράγραφος μόνη της μπορεί να είναι λογική, μπορεί να ξεκινάει από μια καλή πρόθεση, αλλά όλα μαζί δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή τι, επιδιώκουμε μια ομοσπονδιακή ένωση. Τελικά ναι ή όχι. Και πού είναι το όριο. Πώς θα την οριοθετήσουμε αυτή τη ζώνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα σήμερα, αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί τελικά. Εμείς έχουμε μια συμφωνία για τα ευρωμόλογα και το Δεκέμβρη νομίζω ορίσαμε την προθεσμία, πρέπει να την Η δική μου πολιτική ομάδα θα έχει κάποια προβλήματα με αυτό το θέμα ως προς τη διατύπωση. Ε, για την δημοσιονομική εναρμόνιση, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, εκθέσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι εννοούμε ακριβώς. Το CCTB ε, συμφωνούμε. Ξέρουμε ότι πολλοί έχουν ενδιασμούς. Τώρα, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ταμείο, τα χρέη, οι οργανισμοί αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, για όλα αυτά τα θέματα περνάμε ένα, νόημα, ένα μήνυμα συγγνώμη, σήμερα με τη σημερινή έκθεση, αλλά δεν ξέρω αν είναι το σωστό. Η χρηματοπιστωτική εποπτεία. Επ' αυτού κανένα πρόβλημα. Για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ίσω κάποια μικρά προβλήματα και με τη διατύπωση, αλλά τελικά έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή λύση. Η, Ευρωπαϊκή, η στρατηγική 2020 όπως έχει πει επανειλημμένο ο πρόεδρός μας, χρειαζόμαστε περισσότερο μόντι εδώ πέρα. Παγκόσμιες ε, ε, ανισορροπίες. Νομίζω ότι θα γίνουμε πιο υπεύθυνοι με την στρατηγική ε, ε, που θα ακολουθήσει τελικά το G20. θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας κάνετε πιο συγκεκριμένες ε, ε, προτάσεις ε, για αυτό το Συμβούλιο Οικονομικής Ασφάλειας. Αυτή είναι η φρασιολογία του ΟΗΕ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείτε. Τώρα για κάποιες επιμέρους παραγράφους έχω παρατηρήσεις να κάνω, αλλά δεν θα τις αναφέρω τώρα. Ήθελα μόνο να σας κάνω μια ερώτηση για την παιδεία. Αυτή η παράγραφος 47 ενέχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα μπορούσατε όμως να την αναπτύξετε λίγο παραπάνω. Πολλές χώρες μέσα στην Ένωση έχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της παιδείας. Ε, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ποιότητα, παραδείγματος χάρη, της παιδείας. Άλλες πάλι χώρες, όπως η Φινλανδία, έχουν πολύ καλές επιδόσεις. με τις ε, μελέτες πίσω που το καταδεικνύουν αυτό ότι δουλεύει πολύ καλά το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας. Έχω όμως την εντύπωση ότι τελικά ε, προσπαθούμε την ευθύνη να τη μετατοπίσουμε από την εθνική ε, κονίστρα στην ευρωπαϊκή θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε μία προστιθέμενη αξία αν επιδιώξουμε αναβάθμιση της παιδείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς ποια ήταν η πρόθεσή σας, να ε, εξηγήσετε λίγο το περιεχόμενο της παραγράφου 47. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το σύμφωνο EuroSyn. Είναι μια ορολογιακή βόμβα, ουσιαστικά δεν ε, θορυβήθηκα τόσο πολύ με τον τρόπο με τον οποίο το προτείνετε. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε ε, την πρότασή σας ε, και τα πιθανά αποτελέσματά της. Δεν είναι τόσο σημαντική διαδικασία. Μπορώ να συμφωνήσω για την κοινοτική μέθοδο, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Υπάρχουν τέσσερις χώρες που είναι εκτός. Η Βρετανία ποτέ δεν πρόκειται να μπει στη ζώνη ευρώ. Η Ουγγαρία και κάποιες άλλες χώρες και η δικιά μου η χώρα. Δεν συμμετέχουν. Αυτό είναι καταστροφικό για την λειτουργία της Ένωσης. Ποιο... Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ωραία. Το επόμενο ποιο θα είναι. Διαβάζοντας τον τύπο το Σαββατοκύριακο, τον ε, Βρετανικό τύπο συγκεκριμένα, βλέπω ότι όλοι επικροτούν τις εξελίξεις. Πάρα πολύ ωραία, ένα, ένα πρώτο βήμα, μπορούμε να φύγουμε από την Ένωση και να πάμε να προσχωρήσουμε σε κάποια άλλη Ένωση. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε αυτό μέσα στην έκθεσή μας ότι αυτό θα μπορούσε να πλήξει την Ένωση, να παρεμποδίσει την λειτουργία της και βλέποντας τα όσα έχουν συμβεί τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες και ερχόμενος από μια χώρα όπου η αντιπολίτευση στη Βουλή, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, αντιτάχθηκε στην κυβέρνηση και άρα δεν έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της η κυβέρνησή μας για το σύμφωνο Eurosyn. Κλείνει η παρένθεση. Αυτό λοιπόν, αυτή η τάση είναι αρνητική, διότι έτσι μπορεί να διευρυνθεί αυτό το χάσμα, η διχογνωμία που επικράτει στην Ένωση. Προσπαθούν όλοι να βρουν μία λύση, αλλά ο διχασμός είναι βαθύς και νομίζω ότι θα διωγκωθούν περαιτέρω τα προβλήματα. Κυρία Μπερές, ε, νομίζω θα, θα συμφωνήσουμε στο τέλος, αλλά αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ο Πασκάλ, σε ό,τι αφορά τα εισαγωγικά του Αλεσμίτ, συμφωνώ για τη δουλειά της ε, Περβάνς. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με το όραμα που προτείνεται. Εγώ σύντομα θα αναφερθώ στο δέκατο πολύ σημεία, όπου είτε διαφωνούμε είτε έχουμε ερωτήσεις. Δεν θα σας δώσω τη γενική θεώρηση, την κοσμοθεωρία μου ή την κατάσταση του κόσμου, συλλήβδιν, απλώς ε, κάποια πιο επιμέρους ε, σημεία για την έκθεση το πλαίσιο τώρα, δηλαδή στις αιτιολογικές σκέψεις από το άρθρο μέχρι το εφλατινικό, Ακριβώς μιλώντας για θεώρηση αυτή του κόσμου, νομίζω ότι λείπουν κάποια βασικά στοιχεία, κλειδιά, ε, για τα οποία είναι ευρία η συνένεση. Και είναι στοιχεία που έχουν σημασία για το υπόλοιπο της έκθεσης. Το πρώτο που δεν βλέπω και μου λείπει είναι αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία. Μίλησαν πολύ για σας. Δεν είναι μια έκθεση για την ενεργειακή πολιτική μεν, Πριν όμως είναι αρκετά σοβαρά και βαριά αυτά που συνέβησαν και μεγάλη η ε, καμπή ε, στην αντίληψη που έχουμε για αυτά τα πράγματα που έχει και μακροοικονομική επίπτωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στις αιτιολογικές σκέψεις αυτό. Δεύτερον, πληθωρισμός. από τη... τότε που βγήκε το πρώτο τμήμα, πώς να το πω, η πρώτη εκδοχή, εν πάση περιπτώσει, της έκθεσης και μετά, είδαμε ένα νέο οικονομικό φαινόμενο που είναι η αύξηση του πληθωρισμού και πολλοί κεντρικοί τραπεζίτες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική το συζητούν. Θα πρέπει πολύ περισσότερο να το λαμβάνουμε υπόψη από ό,τι σήμερα που δεν τον αναφέρουμε καθόλου. Θα έχει όμως σημαντικές επιπτώσεις αυτό και στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ένα τρίτο που μου λείπει από την έκθεση, και πολύ αναφερθήκατε στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που στην αρχή ήταν χρηματοπιστωτική κρίση, μετά έγινε οικονομική, πολιτική και κοινωνική το 2010, 2009 και 10 μάλιστα, τώρα είναι πολιτική κρίση. Το είπαν ε, επανειλημμένα πολλοί από εσά. Τώρα έχουμε ενώπιό μας ένα πραγματικό πρόβλημα δυνατότητας αποδοχής ορισμένων πολιτικών που ασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις κοινωνίες, από τα έθνη κράτη, από τους λαούς. Είναι ένα ζήτημα αυτό ε, να το αντιληφθούν, να το αποδεχθούν και να ε, ασκήσουν τις πολιτικές ε, κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν πολιτική πλέον η κρίση και θα πρέπει να προβάλλεται περισσότερο στην έκθεση. Ένα τέταρτο στοιχείο που μου λείπει. Τελικά, καμία από τις διαρθρωτικές αιτίε, ε, τις οποίες με ανέφερε η υπερβάνσα, αλλά δεν τις έβαλε στην έκθεση, καμία από τις βασικές διαρθρωτικές αιτίε που οδήγησαν στην κρίση δεν έχει λυθεί σήμερα. Οι παγκόσμιες ανισορροπίες ε, και στην Ευρώπη και στο ε, παντού υπάρχουν, μακροοικονομικά, ε, τα χρέη των τραπεζών επίσης και μεταφράστηκαν σε κρατικά χρέη γιατί ε, τους πέταξαν τον μπαλάκι και το ανέλαβαν οι χώρες τώρα και είναι εκεί που βρίσκονται. Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί, συγγνώμη. Και ένα τελευταίο. Είναι η αύξηση του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς στη Γαλλία, όπως γνωρίζουμε όλοι, αλλά και στη Φιλανδία, όπου επίκυνται εκλογέ. Ξέρουμε ότι είναι και μία απειλή που επικρέμεται επί του Συμφώνου για το Ευρώ και βλέπουμε μετά την πολιτική κρίση ακριβώς ε, η αδυναμία να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση συνδέεται με την αύξηση των λαϊκισμών και αυτό καλό θα ήταν να το αναφέραμε και στις αιτιολογικές σκέψεις. Έρχομαι τώρα στο διατακτικό. Στη ε, παράγραφο 4 και 5 νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο. Ίσως κάνω κάποια τροπολογία εκεί θα δω. Αν χρειαστεί, αν διατύπωση ή και ουσία. Για να επιμείνουμε, λέω, στις συμμετρικές προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε. Τι εννοώ τα ελλείμματα των μεν στην Ευρωζώνη, τα εμπορικά, είναι πλεονάσματα των δε και τούμπαλιν τα πλεονάσματα του ενός είναι τα ελλείμματα του άλλου. Αν θέλουμε να έχουμε μια αντίληψη Ευρωπαίων και όχι απλώς Ελλήνων, Γερμανών, Ολλανδών και τα λοιπά ο καθένας στη χώρα του, θα πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι το ίδιο νόμισμα και έχει δύο όψεις. Τα πλεονάσματα του ενός είναι τα ελλείμματα του άλλου. Ε, αυτή είναι λοιπόν η προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, το ότι βλέπουμε συνολικά την κατάσταση. Για την παράγραφο 5 η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δυνατότητα αποδοχής ακριβώς από τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς των πολιτικών λιτότητας ή δημοσιονομικής εξυγίανσης, για να το πω έτσι με όρους ουδέτερους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και μία φορολογική πτυχή, δημοσιονομική πτυχή. Δηλαδή, αν θέλουμε να μειώσουμε το έλλειμμα, Βεβαίω να περιορίσουμε κάποιε δαπάνε, αν γίνεται, αλλά ταυτόχρονα και οπωσδήποτε και με την ίδια προτεραιότητα να αυξήσουμε τα έσοδα να έχουν τα κράτη-μέλη ε, περιθώρια χειρισμών για να μαζεύουν φόρους και έσοδα που σήμερα δεν μπορούν. Και αυτό είναι στο ίδιο πακέτο δεν μπορούμε να φέρουμε μόνο τους φόρους χωρίς τις δαπάνες, γιατί έτσι χάνουμε κάποιες οικονομίες που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, αλλά δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στο σφίξιμο της ζώνης. Πρέπει να μιλάμε και για ε, τη συλλογή των εσόδων ε, ταυτόχρονα. Λοιπόν, στην παράγραφο 5 θα το έβαζα εγώ. Τώρα δεν είναι θέμα να κάνω μια τροπολογία, είναι ουσίας. Συμφωνούμε να μπει αυτό, να έχουμε ε, μεταξύ μας αυτή τη συμβαστική πρόταση. Ε, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ταμείο. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό και πώς συνδέεται με την, Εθνική Τράπεζα, με την Κεντρική Τράπεζα. Το ρώτησε και ο Όλε Σμιτ. Και στο κεφάλαιο 4 για την ε, ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα ή την εφορία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την αυριανή οικονομία. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ικανότητα που θα έχει η Ένωση να έχει αηφόρο οικονομικό μοντέλο, δηλαδή λιγότερο από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου να ε, αναπτύσσει πράσινες τεχνολογίες, που να είναι ηγετική δύναμη, εν πάση περιπτώσει να στέκει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτή είναι η δική μας θεώρηση και πιστεύουμε ότι και άλλοι συμμερίζονται δεν είναι αντιφατικέ έννοιε η ανταγωνιστική Ευρώπη με την βιώσιμη και αηφόρα οικονομία. Είναι αλληλένδετα, συμπληρωματικά και ε, όρος του, ε, το ένα του άλλου. Για να μην δίνουμε την εντύπωση ότι είναι δύο οι δρόμοι και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ποιον θα ακολουθήσουμε. Στην παράγραφο τώρα 35 έχω μια ερώτηση. Πώς συνδέεται η ενεργειακή πολιτική με την εσωτερική αγορά, γιατί είναι μια κοινή παράγραφος που καλύπτει δύο διαφορετικές πολιτικές και δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Δεν μπορούν να μπουν στην ίδια παράγραφο 35 και σχεδόν τελείωσα. Σχεδόν λέω. Α, στο 57. Το είπε και όλοι προηγουμένως. Νομίζω ότι δύσκολα πραγματικά μπορούμε σήμερα να ζητούμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και βάθυνση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον τρόπο της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν βλέπω να το έχετε καλύψει επαρκώς σήμερα. Δεν υπάρχει βούληση μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών να έχουμε πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση χωρίς παράλληλα ποιοτικό άλμα στη λειτουργία ε, της υπευθυνότητα, της λογοδοσίας παντού, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε όλα τους τα επίπεδα. Και βέβαια είμαστε υπέρ μιας οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και βαθιάς, αλλά αυτή δεν πρόκειται να γίνει στα πλαίσια της σημερινής λειτουργίας των σημερινών θεσμικών οργάνων και θα πρέπει και αυτό να αναφερθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πασκάλ. Τελευταίο συντονιστής, ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συγγήτρια, μετέχοντας εδώ και 1,5 χρόνο στις διαδικασίες της Επιτροπής, οφείλω να σας πω ότι κατονοώ τη δυσκολία που έχει και η συγγήτρια και εμείς και πολύ περισσότερο στη διαδικασία να συντάξουμε το τελικό κείμενο. Ποια είναι η δυσκολία μας. Έχουμε τους περιορισμούς της ενδιάμεσης έκθεσης, όπου σε βασικά ερωτήματα απαντάει κατά διαφορετικό τρόπο από αυτό που θα ήθελα, αλλά και ταυτόχρονα λόγω του συγκεκριμένου συσχετισμού έχουμε ορισμένα ιδεολογικά πολιτικά κλισέ, θέλουμε να ερμηνεύσουμε πράγματα που δεν ερμηνεύονται με αυτά και πάμε να τα κλείσουμε σε ένα κείμενο που στην πράξη είναι διάτριτο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου. Πέρα από τις προθέσεις μας. Πέρα από τις προθέσεις μας. Και με αυτή την έννοια, ε, αγαπητέ Πρόεδρε, επιτρέψτε μου και αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια πρόταση που έχει και συμβολικό χαρακτήρα ίσως. Επειδή και η συγγήτρια ξεκίνησε την παρουσίαση της έκθεσής της, αλλά και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν ότι η κρίση δεν έχει περάσει. Ορισμένες από τις βασικές αιτίες, αυτές που κατέγραφε το κείμενο, δεν έχουν θεραπευθεί. Προτείνω να ζητήσουμε την παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής μας. Και δεν το λέω καθόλου αστιβόμενος. Θυμάμαι, ότι η παράταση για ένα ακόμα χρόνο, εκτός των άλλων λόγων, έγινε για να μην δώσουμε το μήνυμα ότι η κρίση πέρασε. Έτσι δεν είναι. Όσο θα υπάρχει κρίση, και πολύ φοβούμε θα υπάρχει με διάφορες μορφές, τότε η Επιτροπή μας, λέω εγώ, να προτείνουμε να συνεχίσει τη λειτουργία, ενδεχομένως και γίνει μόνιμη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτές είναι οι δικές μου προβλέψεις, και ναι, ενδεχομένως, με, την, με, την, με την ελπίδα με την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία, μήπως, μήπως ορισμένες από τις προτάσεις μας, ορισμένες επιμέρους προτάσεις, στις οποίες μπορώ να συμφωνήσω και εγώ, γίνονται κάποτε δεκτές. Μήπως ορισμένες από αυτές τις προτάσεις εφαρμοστούν εν μέρη. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση έχει και αυτή το στοιχείο μιας άλλης πρότασης. Επειδή και ο αγαπητός Πρόεδρος και ο αγαπητός φίλος ο κύριος Σμιθ σχολίασαν ε, ε, κατέθεσαν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στην Ελλάδα. Θα έλεγα στο φίλο τον κύριο Σμιτ, απογοητεύτηκε λέει γιατί οι πολίτες στην Ελλάδα του έδωσαν την εντύπωση ότι δεν θέλουν να αλλάξουν, χωρίς παρεξήγηση. Αν πάρουμε σαν κριτήριο ότι η χώρα του και κατ' επέκταση οι πολίτες δεν μπαίνουν τόσο καιρό στο ευρώ, αν πάρουμε υπόψη ότι η, η, η Σουηδία δεν δέχεται να μπει στους μη, τα μη μέλη του ευρώ στο σύμφωνο του ευρώ, πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι Σουηδοί δεν θέλουν να αλλάξουν μυαλά, δεν θέλουν να γίνουν καλοί, δεν θέλουν να πειθαρχήσουν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και δεύτερο, αγαπητοί συνάδελφοι, είπε ο Πρόεδρος, και έτσι είναι, αυτή είναι η εικόνα, δεν είναι διαφορετικό, υπάρχει μια πολιτική διαμάχη στην, στην Ελλάδα. Δεν, θεωρού, δεν θεωρείται ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι εθνικό πρόγραμμα. Και έτσι είναι τα πράγματα. Δείτε και την Πορτογαλία και μην το θεωρείτε ξεχωριστό φαινόμενο. Είναι πολιτικές επιλογές. Δεν είναι αναδύρυτη, αδύρυτη οικονομική ανάγκη αυτό που γίνεται. Μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Και να ήταν και πιο αποτελεσματικό. Επομένως, όσο περνάνε και εισπράττουν οι πολίτες πολιτικές τέτοιες, δεν μπορούν να το εκλαμβάνουν ως εθνική πολιτική. Δηλαδή θα μπορούσε να πει το κείμενό μας, θα μπορούσε να είχε ε, δεν ξέρω αν είναι στα αρμοδιότητέ μα, μια αξιολόγηση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από συγκεκριμένε χώρε για να βγούμε από την κρίση. Και να δούμε ότι δεν βγαίνει. Απλώ ανακυκλώνεται η κρίση. Όλο αυτό λοιπόν το σκεπτικό για να μην σα κουράζω καταλήγει στο εξή. Στην εξή πρόταση. Για να καταλάβουμε αν οι Έλληνε θέλουν να αλλάξουν. Αν οι Σουηδοί κάνουν κακό που είναι εκτό ευρώ και δεν συμφωνήσαν να είναι στην ομάδα αυτών των μη χωρών μελών του ευρώ. Η πρόταση τη ε, της δικής μας Επιτροπής πρέπει να συμπληρώνεται και επειδή σωστά ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί την νομιμοποίησή της από τις δημοκρατικές αρχές, να ζητήσουμε να διενεργηθούν δημοψηφίσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Συμφώνου για το Ευρώ. Γιατί το αποφεύγουμε. Ποιος ξέρουμε αν το εγκρίνει ή όχι. Διότι περνώ σε μια επιμέρους παρατήρηση που περιλαμβάνεται στο κείμενο. Αν θεωρούμε ότι με το σύμφωνο για το ευρώ, που από ό,τι φάνηκε υπερκάλυψε το πακέτο που συζητάει εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπαμε να τελειώσουμε στο 2000 τον Ιούνιο για την οικονομική διακυβέρνηση, αν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα βήμα για περαιτέρω οικονομική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, φοβούμε κύριοι συνάδελφοι ότι πάμε σε μια Ευρώπη πιο συντηρητική, πιο αντιδημοκρατική και πιο αντικοινωνική. Έτσι ένα όραμα που θα είχε κανείς, το έχω κι εγώ, για μια ενιαία πολιτική Ευρώπη, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά, αυτό όλο και περισσότερο αμαυρώνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάρει δημοκρατική νομιμοποίηση αυτό το βήμα και αυτή είναι η δεύτερη μου πρόταση. Δημοψήφισμα, λοιπόν, α το προτείνουμε και η Επιτροπή, γιατί είναι όχι, για να υιοθετηθεί ή όχι από τι χώρε και από του ευρωπαϊκού λαού το σύμφωνο για το ευρώ, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, ορισμένε επιμέρου παρατηρήσει, διότι το διάβασα το κείμενο και αξίζει τον κόπο να μπούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις. Στην αρχική, στην αρχική σελίδα, στο σκεπτικό Β, νομίζω ότι δεν αποδίδεται καλά η, η εξεγέρση στον αραβικό κόσμο. Είναι μια παρεξηγήσιμη τοποθέτηση κατά τη γνώμη μου. Το συνδέει κατά μία έννοια με την οικονομική σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι βάζει το θέμα ότι είναι μια υπενθύμηση των αρχών της δημοκρατίας. Οι εξεγέρσεις κατά τη γνώμη μου έχουν έντονα κοινωνικό χαρακτήρα και η έκφραση αυτή νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστική να το πούμε ότι εμπορικές ανταλλαγές ας πούμε δεν πήγαν καλά ας πούμε της Αιγύπτου και τη Σουηδίας πάλι θα α, αναφερθώ στο φίλο μου το Σμιτ και αυτό ήταν το πρόβλημα ας πούμε που είχαμε τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο και εκεί. Ε, τώρα, ε, έχω ξαναπεί για το χρέος και ορισμένα φαινόμενα τα εξηγεί. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, έχουμε φτάσει το αποτέλεσμα να θεωρείται αιτία, η κρίση χρέους. Θα άξιζε τον κόπο, ίσω και για αυτό το λόγο, μια παράταση τη θητείας τη Επιτροπής μα ή και με τη συνδρομή άλλων επιτροπών, να εξεταστούν τα ποιοτικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, του χρέου, ιδιαίτερα σε χώρε που εμφανίζουν υψηλό χρέο. Αν προσπάθησα να δω, υπάρχουν διαφορέ. Αλλού είναι μεγάλο το δημόσιο χρέο, αλλού είναι μεγαλύτερο το ιδιωτικό χρέο. Και εννοώ τι χώρε που εμφανίζουν χρέο, δεν εννοώ τι άλλε, τι αμόλυντε και προ το παρόν χωρί τέτοια προβλήματα αλλού είναι μεγαλύτερο το εσωτερικό χρέος, αλλού είναι μικρότερο το εσωτερικό χρέος, που σημαίνει ότι πρέπει να δεις ποιες είναι οι πιο συγκεκριμένες ευθύνες του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού για την κρίση χρέους που εμφανίζεται κάθε χώρα και νομίζω ότι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα βοηθούσαν στο να δούμε καλύτερα ορισμένα πράγματα. Θέλω να σας πω ότι η ομάδα μου διαφωνεί με τη συνταγματική αναθεώρηση και αυτό το μηχανισμό σταθεροποίησης και διαφωνούμε πάρα ε, κάθετα θα έλεγε κανείς και με τη, ε, ε πούμε κατηγορηματικά και με τη διαδικασία που φαίνεται ότι ακολουθείται με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 48 και όχι με τη συνήθη διαδικασία. Διότι αυτή η αναθεώρηση ουσιαστικά δίνει αρμοδιότητες στην Επιτροπή, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τροποποίηση τις συνθήκης και απαιτεί συνήθη διαδικασία, δηλαδή ε, συνέλευση και τη διαδικασία που προβλέπει το 48-2 αν δεν κάνω λάθος, ενώ με τη διαδικασία που γίνεται, νομίζω ότι γίνεται παραβίαση των συνθήκων και αποδίδονται στην ε, Επιτροπή ε, ε, συνθήκες που, αρμοδιότητες συγγνώμη, που, δεν έχουν, που δεν έχει. Άλλωστε, η ποιοτική διαφορά μεταξύ τη απλοποιημένη και τη συνήθους διαδικασία όπω την έχω αντιληφθεί από τη μελέτη του σχετικού άρθρου, είναι αυτό ακριβώ, αν αποδίδονται ή όχι ευθύνε. Δεν θέλω να σα κουράσω περισσότερο, υπάρχει ένα θέμα στι παγκόσμιε ανισορροπίε όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Εδώ δεν αναφερόμαστε σε αυτή την, ε, δυστυχώς, τη διαδικασία που ξεκίνησε με τη δεύτερη θητεία ιδιαίτερα της νέας Κομισιόν με το άνοιγμα του δρόμου για τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη, με συνεχείς αποφάσεις. Και εδώ είναι επιτακτικό να τεθεί το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, να στηριχτεί το αγροτικό εισόδημα και να γίνει μια αναθεώρηση της ε, ε κοινή αγροτικής πολιτικής. Γρήγορα, άλλη μια φορά στο επάρατο, ε, ε, το στο κακόφημο Διεθνές Ρομισματικό Ταμείο. Δεν το μπορώ <laughs> να σας το πω έτσι. Όπου έχει πάει είναι καταστροφή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αναγνωρίζουμε. Βέβαια το ξεκίνησε η χώρα μου, θα έλεγα και εγώ τώρα, όπως αποδείχθηκε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργό έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωζώνη. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα το βάζουμε να συνδιαμορφώνει τι πολιτικέ. Και να το δεχόμαστε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κάνουμε προτάσει που να περιλαμβάνει και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δεν θα το ήθελα, αλλά εν περιπτώσει δεν θα κουραστώ να λέω την άποψή μου, έστω και αν είναι ψηφούσα, Τελειώνω γρήγορα, αγαπητέ Πρόεδρε. Από εκεί και πέρα ε, για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική 2020 που περιλαμβάνεται σε αρκετά σημεία, θεωρώ. Μ, πώς να σας το πω. Ε, Συσίφιο το έργο, ο γνωστό μύθο του Συσίφου, υπήρχε μια πέτρα, την έφτανε μέχρι πάνω και όταν έφτανε πάνω το έφευγε. Δηλαδή δημοσιονομική προσαρμογή και αναπτυξιακή πολιτική δεν <laughs> Κατά τη γνώμη μου ε, και επομένω η ρητορία εκεί δεν μα βγάζει σε τίποτα. Τέλο, μια πινελιά ακόμα στο θέμα τη εκπαίδευση και θα σα ε, ευχαριστήσω για την ανοχή σα. αυτή η λογική που είναι κυρίαρχη να υπαγορεύεται και να υπαγάγεται η εκπαίδευση τη ανάγκη αγορά δεν νομίζω θα μας βγάλει υψηλός, υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό, αλλά μάλλον ένα ευέλικτο δυναμικό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά όπως βλέπετε τώρα όλα μας γίνονται κατά το κριτήριο για τις επιχειρήσεις να σταματήσουν να είναι ανήσυχες οι αγορές. Με αυτές τις προτεραιότητες φυσικά γίνονται αυτές οι προτάσεις. Τώρα, τελειώνω. Δεν θα το ψηφίσουμε από ό,τι φαίνεται το κείμενο και λέω από ό,τι φαίνεται γιατί δεν έχω κάνει συνεννόηση και με τα άλλα μέλη τη ομάδας. Στα σημεία που ανέφερα και άλλα που έχουν αναφερθεί θα καταθέσουμε λίγες τροπολογίες, γιατί δεν αξίζει βέβαια να ταλαιπωρούμε την εισηγήτρια με άλλες τροπολογίες. Θα καταθέσουμε τροπολογίες στα βασικά θέματα και θα συμμετέχουμε στη συζήτηση. Ευχόμαι ότι κάποια στιγμή ενδεχομένω αυτά που λέω εγώ ή που θα πούμε να γίνουν κοινώ παραδεκτά και να τα παλέψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ, Νικό. Η ΣΥΡΠΑ τώρα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, ε, πολύ καλή δουλειά της, πολύ σχολαστική. Είναι ισοσκελισμένη η πρότασή σου και ναι, έχει στοιχεία που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη και γίνεται συγκερασμός πολιτικών απόψεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες αλλά η ποσότητα και η ποιότητα, το περιεχόμενο των τροπολογιών τουλάχιστον ε, θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα, ούτω ώστε να διατηρηθεί η τωρινή δομή και έτσι να εγκριθεί τελικά το σχέδιο έκθεσης. Δεν ε, θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, θα ήθελα όμως να σχολιάσω κάποια ζητήματα που μας ικανοποιούν σε πρώτο λόγο και δεύτερον αυτά που μας προβληματίζουν. Στον πρώτο γύρο Πολλοί μίλησαν για τον έλεγχο του χρέους, ε, για την ευθύνη, για την αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω ότι η διατύπωση είναι καλή, ισορροπημένη για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, ε, προβληματίζομαι πως πρέπει να διευρύνουμε λίγο τη διατύπωση. Γνωρίζω ότι είναι ακαθόδες το θέμα από πολιτική σκοπιάς. και σχετίζεται με κάτι άλλο που αναφέρεται, δηλαδή ε, το πώς συμβαδίζει ο προϋπολογισμός της Ένωσης με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Να σε εξηγήσω τη σκέψη μου. Χρειαζόμαστε την κοινωνική ευθύνη, χρειαζόμαστε κοινωνική ένταξη, χρειαζόμαστε αναπτυξιακά στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να ε, ε, αυξήσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περικοπές στις δαπάνες και στις επιδοτήσεις, στις παροχέ ως προς τις τομεακές πολιτικές, κυνηγιορική πολιτική, πολιτική συνοχής κτλ. Είναι ζήτημα. Θα συνεχίσουμε τη Θα, θα πραγματευτούμε εδώ αυτά τα ζητήματα η κοινωνική ευθύνη, η μελλοντοστραφή πολιτική και οι επενδύσει στο μέλλον είναι τρία πράγματα που συμβαδίζουν, αλλά πρέπει να δείτε και το τι σα επιτρέπει ο προϋπολογισμός σας. Ε, δηλαδή, αν δεν μπορείτε ε, να αυξήσετε τα κονδύλια σα, θα πρέπει να ε, στείλετε άλλε δαπάνε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κατόπιν μιλάτε για την οικονομία που βασίζεται στι γνώσεις και τονίζετε τη σημασία της παιδείας. Προφανέστατα, είναι βασικός, ακρογωνίω λύθο η Τώρα αυτή η συζήτηση αν πρέπει να ε, τοποθετηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο διαφέρουν οι απόψεις. Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουμε θα διαφέρει και η ευθύνη, η λογοδοσία δηλαδή στον τομέα αυτό. Για την αναπτύξη, πολύ καλά τα σχόλιά σας. Και πάλι τίθεται το ζήτημα αν συμβαδίζει ο προπολογισμό Ένωση με του εθνικού προπολογισμού, μικρομεσαίε επιχειρήσει, καινοτομία, όλα αυτά ωραία. Αλλά γιατί ξεχνάμε το venture capital, ε, δηλαδή το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, γιατί ξεχνάμε γενικότερα το ιδιωτικό κεφάλαιο και δεν το συζητούμε από κοινού με την πολιτική καινοτομία. Ε, στην παράγραφο 36 θα ήθελα να πούμε περισσότερα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και ε, για την υποδομή και για τις επενδύσεις ε, που τρέχουν. Δεν μπορείτε δηλαδή να λύνετε τα θέματα ε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ανάπτυξης αποσυνδέοντάς τα από τους πόρους, από την έλλειψη πόρων πιο συγκεκριμένα για τη χρηματοδότησή τους. Βλέπετε τις τιμές των τροφίμων που αυξάνονται Βλέπουμε τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, η... είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε για ενέργεια, για πρώτες ύλες, ε, για, ε, για το καθαρό πόσιμο νερό, για την χρήση της γης, οτιδήποτε, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ μέσα στην έκθεση ε, είναι ή μάλλον να το πω αλλιώ. αναφέρεται μέσα στην έκθεση για, για τον κανονισμό για την χρηματοπιστωτική εποπτεία ότι μόνο κάποια πρώτα βήματα έχουν γίνει και ότι δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα άλλα περαιτέρω βήματα. Ως προς την ε, ισχυρή παγκόσμια προσέγγιση, αυτή την ιδέα που προτείνετε μέσα στην έκθεσή σας, καλή ιδέα είναι αλλά χρειάζεται υψηλότερη φιλοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να λειτουργήσει ως παγκόσμιος παίκτη και να υλοποιηθούν αυτά που προτείνεται στην έκθεση. Ο ρόλος της ομάδας G20, το Συμβούλιο Οικονομικής Ασφάλειας, ε, όλες αυτές οι ιδέες που βλέπουμε στην έκθεσή σας, ε, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Κατόπιν, δύο βασικά ε, πολιτικά ζητήματα που θέλουν να συμπεριληφθούν, να τονιστούν περισσότερο στην εκθεσή σας. Η κοινοτική μέθοδος σε διάφορα σημεία του κειμένου αναφέρεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ένωση. Μήπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε περισσότερο, να εξηγήσουμε τι εννοούμε ακριβώς, αν πρόκειται δηλαδή να συντονίζονται οι εθνικές οικονομικές πολιτικές μέσω ε, της κοινοτικής μεθόδου. Τι σημαίνει αυτό για τη βιωσιμότητα και την αηφορία και άλλα στοιχεία των οικονομικών πολιτικών. Θα σταματήσω εδώ για αυτό το σημείο. Τώρα επανέρχομαι σε σχόλια του Όλε και άλλων. Έχουμε πολιτική κρίση επίσης, ναι ή όχι. Άλλο δύσκολο ζήτημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω απαντήσεις. Ε, φανταστείτε δύο σιαμαία δίδυμα αλλά ε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε τρεις, ε, τρία αδέλφια. Έχουμε την δημοκρατία, έχουμε την ελευθερία και την οικονομία. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν για να μην έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε τις αλλαγές. Αν οι άνθρωποι δεν θέλουν τις αλλαγές δεν μπορείτε να τις επιβάλλετε. Όμως αν ισχύει το αντίθετο... Και τώρα θυμίζουν αυτά που λέω λαϊκισμό. Όταν διαπιστώνεται κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, σκέφτονται οι άνθρωποι, μα είναι λάθος των πολιτικών, δεν μας προστάτευσαν αρκετά. Έχουμε εκχωρήσει υπερβολικά μεγάλη εξουσία σε αυτή την παγκόσμια οικονομία. Έτσι σκέφτονται. Μερικώς αληθεύει αυτή η θεωρία. Παιδεία τώρα δεν είναι θέμα μόνο ανταγωνιστικότητας η παιδεία. Όποια ε, πεφωτισμένη διαδικασία λήψη αποφάσεων και αν ακολουθήσουμε, το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε την, ε, το, πώς έχουν τα πράγματα στην ουσία για να βρούμε μία λύση. Ε, ακούσαμε επίσης ότι πρέπει να τρέχουν οι πολιτικοί ηγέτες και να μην μπορούν να τους παρακολουθήσουν οι άνθρωποι. Μα εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει αυτό με στην Ένωση. Μάλλον το αντίθετο, μάλλον άλλο πρόβλημα έχουμε. Εντάξει, εγώ είμαι από τη Φιλανδία, έχουμε και τις εκλογές, τέλος πάντων και στη Σουηδία πρόσφατα το ίδιο θέμα είχατε. Τι συμβαίνει λοιπόν. προσπαθούν κάποιοι να τρέξουν και να πάρουν την σημαία και να πούνε εγώ είμαι ε, ο ηγέτης. Για φα, πάρτε ένα άλλο παράδειγμα, ένα γιατρό και έναν ασθενή που έχουν ασθενή σχέση και καταλαβαίνει ο ασθενή ότι καλό είναι να πάρει κάποια αναλγητικά γιατί εν πάση περιπτώσει δεν του αρέσει η ιδέα της εγχείρηση και θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι. Τι θα πει ο γιατρός, θα συμφωνήσει με τον ασθενή για να μην ταράξει τον ασθενή και αλλάξει ε, ιατρικό κέντρο που θα είναι, ε, ή να ακολουθήσει άλλη θεραπευτική αγωγή που θα είναι χειρότερη ή θα προσπαθήσει να πείσει τον ασθενή και να το εξηγήσει γιατί μπορεί και να χρειάζεται όντω επέμβαση και δεν χρειάζεται μόνο θεραπευτική αγωγή. Έτσι τίθεται το δίλημα κατά τη γνώμη μου. Καλύτερο θα ήταν να εξηγήσουμε την ε, κοινοτική μέθοδο για να έχουμε, να αποκτήσουμε περισσότερη Ευρώπη. Ε, δεν πρέπει να υποτιμούμε το ζήτημα, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η κρίση είναι μια πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Αλλά γιατί δεν τα καταφέρνουμε. Νομίζω θα έπρεπε να προβληματιστούμε για την πορεία της δημοκρατίας δεδομένων των εξελίξεων. Ευχαριστούμε. Η Λίζα Γιακονσάρη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε ακόμα αυτή την έκθεση για να ξέρουμε και ποιο μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και να είναι σαφέστερο το μήνυμα. Είναι πολλές οι κρίσεις, δεν είναι μία. Κρίση χρέους, κρίση ανταγωνιστικότητας ε, κρίση γενικότερη. Αλλά μπορεί να βρεθεί λύση. Το είπε και η ΣΥΡΠΑ προηγουμένως. Αλλά η μεγαλύτερη κρίση και άλλοι συνάδελφοι είναι η κρίση δημοκρατίας. Το είδα πρόσφατα κι εγώ στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Ο κύριος Παρόσο είναι Πορτογάλος ο ίδιος και δεν κατάφερε να πείσει την ίδια τη χώρα του, ε, τους πολιτικούς της χώρας του για το νόημα που θα είχε μια ε, οικονομική πολιτική. Αν δεν μπορείς να το κάνει ο κύριος Μπαρόσο, ποιος θα το έκανε. Καταλαβαίνω ότι είναι υπεράνω της εθνικής πολιτικής, αλλά ε, βλέπουμε ότι έχουμε έλλειμμα και εκεί. Αν δούμε τι έγινε τώρα για το ευρώ, το περίφημο σύμφωνο για το ευρώ ή ε, Europlus, ξέρω. Το συζητάμε στο κοινοβούλιο και με ποιο τρόπο. Άντε να το έχουμε συζητήσει μία ή δύο φορές το πολύ. Ενώ οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Οι προτάσεις μας κατακλείζουν είναι πολύ δύσκολο καν να παρακολουθεί κανείς όσα λέγονται και γίνονται. Κρίση χρέους τελικά έγινε κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και μένα αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Αυτό που ρώτησε όλοι Σμιτ, τι μήνυμα θέλουμε να δώσουμε με την έκθεση αυτή, τι να βγει, τι θέλουμε, μια Ευρώπη πιο ομόσπονδη, φεντεραλισμό, Αν θέλουμε συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντονισμός σήμερα ονομάζεται διακυβέρνηση, governance. Η εποπτεία των τραπεζών είναι κάτι το ανέφικτο περίπου, γιατί οι τράπεζες είναι παγκόσμιοι ε, πρωταγωνιστές πλέον και διεθνείς ε, οργανισμοί. Ε, δεν μπορεί να γίνει πλέον η εποπτεία των τραπεζών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται είναι ευρωπαϊκή εποπτεία. Και αυτό σημαντικό μήνυμα. Και κάτι άλλο. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει και ο συνάδελφος από την Ελλάδα. Σε αντίθεση με τους λαϊκιστές, οι περισσότεροι από εμά εδώ πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι η λύση, δεν είναι το πρόβλημα. Και η λύση ε, βρίσκεται και... Ε, ασκείται σε διάφορα επίπεδα. Δεν ξέρω ε, εάν μπορούμε σήμερα να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την έκθεση αυτή. Για το, το, το πνεύμα της ε, έκθεσης όμως ε, το καταλαβαίνουμε και ε, αναφέρεται πολύ και στην εκπαίδευση, αλλά όχι με τη στενή έννοια. Εκπαίδευση, παιδεία μπορεί να σημαίνει ικανότητες, δεξιότητες, ανταγωνιστικότητα, μεγάλους στόχους, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να κάνουμε κάτι έχοντας υπόψη μας το κοινό καλό όλων στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να διδαχθούμε και από την κρίση. Τι μάθαμε από την κρίση. Μάθαμε τίποτα. βλέπουμε πάλι οι τράπεζες να μοιράζουν μπόνους και μάλιστα αυξημένα. Μάθαμε τίποτα από την κρίση αυτή. Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια ευφυής προσέγγιση, ένας ευφυής τρόπος ε, αντιμετώπισης και αυτό ε, τονίζουμε την παιδεία. Αν θέλουμε περισσότερη παραγωγή στην Ευρώπη, χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη παιδεία, αλλά και ε, τελικά αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Ναι. Κάτι άλλο που λείπει από την Ευρώπη είναι Ευρωπαίοι διανοούμενοι, στοχαστές. Δεν συμμετέχουν αυτοί ε, στη αναζήτηση της λύσης. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην Περβάνς, λέει ο Πρόεδρος, ε, για να συνοψίσει κάπως ή να απαντήσει κάπως σε όλα τα σχόλια και τις προτάσεις που ακούσαμε. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ μερικά λόγια. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι δεν πέρασε η κρίση. Απλώς αλλάζει χαρακτήρα η κρίση, μεταβάλλεται, τώρα έχει γίνει πολιτική. Και μάλιστα συστημική θα έλεγα, της οικονομίας της αγοράς. Όλο και περισσότερο αυτό το επικρίνουν και το αμφισβητούν οι πολίτες. Να προσθέσουμε ότι που φαίνονται ε, σκόπιμα και χρήσιμα. Βέβαια θα δείξει το μέλλον αν ήταν χρήσιμα και σκόπιμα τα μέτρα αυτά, αλλά δεν αρκούν. Διότι η συμπεριφορά δεν αλλάζει, οι συμπεριφορές του κόσμου, το mindset, η νοοτροπία, η συμπεριφορά, η αντίληψη που προκάλεσε σε κάποιο βαθμό και την κρίση. Δεν άλλαξε, τουλάχιστον δεν άλλαξε ριζικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί αν όλες αυτές οι προτάσεις που κάνουμε και ήδη εφαρμόζουμε όλες αυτές οι ιστορίες της ρύθμισης, αν πραγματικά βρίσκουν το στόχο τους. Γιατί αν δεν αλλάζει ο κόσμος τακτική, οι, οι φορείς, οι ενεχόμενοι, τι να τους κάνουν μερικούς επιπλέον νόμους ή ρυθμίσεις ε, για την εφαρμογή τους αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός και ευρώ δεν εννοώ το νόμισμα αλλά την Ευρώπη. Ευρωσκεπτικισμός, ε, επιφυλακτικότητα και αρνητική στάση απέναντι στην Ευρώπη την ίδια. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αν θέλουμε να τη διαμορφώσουμε μακροπρόθεσμα ε, δημιουργικά, να καταστρέψουμε αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό. Γιατί εμείς θέλουμε την Ευρώπη των πολιτών. Και όταν λέμε ότι θέλουμε περισσότερο Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη και συμφωνούμε εδώ, ε, θα πρέπει να πούμε τι θα πρέπει να δώσουμε πίσω στους πολίτες. Γιατί αν τραβάμε υπερβολικά το πάπλωμα προς την Ευρώπη ή τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να δώσουμε κάτι και στους πολίτες. Γιατί τα συγκεντρώνουμε όλα προς τα δω. Αυτό λείπει και από την έκθεση. Θα έχουμε και μία προσφορά στους πολίτες. Ποιοι είναι οι τομεί που είμαστε πρόθυμοι να πούμε ότι ε, δεν χρειάζεται αυτό να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το επιστρέφουμε σε επίπεδο εθνικό και ενίοτε περιφερειακό. Εδώ έχουμε μια μεγάλη σύγκρουση. Από τη μια θέλουμε να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και από την άλλη βλέπουμε ότι η αρχή της δημοκρατίας ε, επιβάλλει να λαμβάνονται οι αποφάσεις κοντά στο πολίτη. Αυτό είναι μια αντίφαση. Πώς θα ευαθύνεις από μια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λαμβάνοντας τις αποφάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και κοντά στον πολίτη. Εκεί θα κληθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και ένα τελευταίο. Μπορούμε να πούμε, έτσι με ίσχυε τη συνείδησή μας ότι το ευρώ δεν είναι μόνο ένα νόμισμα, αλλά είναι και ένα πολιτικό εγχείρημα και σχέδιο. Και εφόσον είναι πολιτικό εγχείρημα και σχέδιο, να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτό, μακροπρόθεσμα τελικά θέτει αυτόν εκτός Ευρώπης. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που μακροπρόθεσμα, δεν λέω τα επόμενα δύο-τρία χρόνια, μακροπρόθεσμα δεν θέλει να εστερνιστεί αυτό το πολιτικό όραμα που λέγεται ευρώ, τότε θέτει τον εαυτό του εκτός ενώσεως και να πάει να γίνει, ξέρω εγώ, μέλος του ΕΟΧ, Λίχτενστάιν, Νορβηγία, συνδεδεμένο μέλος, εν πάση περιπτώσει να μην είναι πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα το πω και στους Βρετανούς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό το σθένος να το πούμε στην Επιτροπή μας, να πούμε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή τι είναι. Και δεν μιλάω για τη Σουηδία, γιατί γνωρίζω ότι η Σουηδία κάποια στιγμή θέλει να μπει. Βασικά όλοι θέλουμε, ξέρεις, στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, στη Δανία Εξαρτάται αν θα μπει πρώτη η Σουηδία ή δεν ξέρω κάποια άλλα βορειοευρωπαϊκά κράτη ή τα νέα κράτη-μέλη από την Ανατολική Ευρώπη. Τώρα έχουμε την εξή κατάσταση λοιπόν. Και αυτό είναι νέο. Παίρνουμε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι υποχρεωμένα να συμφωνήσουν σε αυτές κράτη που αρνούνται να μπουν στο σχέδιο του ευρώ. Ε, και αυτό δεν είναι δίκαιο έχουν ένα μοχλό θα έλεγα πίεση στα χέρια τους και τους επιτρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή, δυσανάλογα μεγάλη επιρροή. Περβάς, όπως πάντα έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω Αλλά καταρχήν τρεις αρχικές παρατηρήσεις. Πρώτο, το είπα στην εισαγωγή μου, αλλά το ανέφεραν πολλοί στις τοποθετήσεις τους, οπότε και εγώ επανέρχομαι. Αυτοί που είχαν αμφιβολίες για το εύρος της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, αλλά και στο εύρος των απαντήσεων που πρέπει να δοθούν για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, δυστυχώς Όλοι αυτοί διαψεύδονται. Και εγώ χαίρομαι που συλλογικά πήραμε την απόφαση να παρατείνουμε την εντολή. Εγώ προτείνω σχετικά με την εντολή να μην την ξεκινήσουμε τη συζήτηση ευθύ αμέσως πρέπει να μετράμε εμείς τη δυνατότητα παρέμβασης μιας επιτροπής σαν τη δική μας. Είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της εντολής μας ορισμένες ομάδες ήταν λίγο πολύ παρούσες. Οι λύσεις ε, που δώσαμε στην πρώτη έκθεση είναι είναι ακόμη επίκαιρες γιατί σίγουρα δεν διαψεύθηκαν αλλά δεν είναι όμως και λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν αύριο, είναι μακροπρόθεσμες λύσεις. Πρέπει κατά συνέπεια ανανεώνοντας την εντολή μας να δούμε και την αποτελεσματικότητα του μηνύματός μας. Και για να έχει και νόημα η παράταση της εντολής μιας επιτροπής αντιδική μας, πρέπει να είναι πραγματικά υπόθεση όλου του Κοινοβουλίου. Να είναι δηλαδή κινητοποιημένο το Κοινοβούλιο. για την ύπαρξη αυτής της Επιτροπής και την δυνατότητα μοχλού που έχει. Εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε άμα είναι για να ξαναπούμε τα ίδια πράγματα που λέγαμε, ε, που είπαμε και παλιά, και ούτε μόνο να υπάρχουμε για να είμαστε δέκα βουλευτές σε μια γωνιά, χωρίς να αντικατοπτρίζεται ο γενικός προσανατολισμός του οργάνου. Και φυσικά δεν έχουμε και κανένα λόγο ύπαρξης άμα δεν καταλήγουμε και σε νεοτεριστικές λύσεις για την πραγματικότητα της κρίσης. Ορισμένοι συνάδελφοι το είπαν να υπάρξουν τροπολογίες για τις δύο τελευταίες εξελίξεις. να γίνουν τροπολογίες για αυτά τα νέα σημεία τα οποία έχουν προκύψει και μπορεί να λένε, που μπορεί να λένε ότι δεν μπορούμε εμείς να θεωρούμε ότι τα πάντα εδώ λειτουργούν σε αλληλοσύνδεση. Αλλά δείτε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αραβική Άνοιξη Το τι έγινε στην Τινησία α πούμε δεν είναι, είναι πράγματα καινούργια που γεννιούνται από μέσα. Δεν είναι οι Γάλλοι Μαουικοί οι οποίοι ξαφνικά να κάνουν επανάσταση στην Τινησία. Είναι η γενικότερη απελπισία που οδήγησε σε αυτές τις αλλαγές στην Τινησία. Η αδυναμία ενσωμάτωσης αυτής της χώρας στους παγκόσμιους μηχανισμούς. Οι στρατηγικές των πολυεθνικών δεν συνέβαλαν στην δημιουργία ε, αϊφόρων θέσεων εργασίας, δεν ήταν κατάλληλες για να παίξουν ένα θετικό ρόλο σε αυτές τις χώρες. Οι πλούσιοι αυτών των χωρών ε, αντί να επενδύουν επί τόπου που βγάζανε τα πετρελοκέρδη τους ε, στο εξωτερικό, τέλος πάντων όλα αυτά παγκόσμια ισχύουν, έχουν επιπτώσεις στον οικονομικό, κοινωνικό τομέα. Απ' την άλλη μεριά πάλι έχουμε στην ε, Ιαπωνία πάλι ένα καπιτολιστικό φαινόμενο, μία τρέλα δηλαδή του να, κερ... να χτίζει κανείς πυρηνικά εργοστάσια πάνω σε ένα σεισμικό ρήγμα. Δηλαδή αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν και για την πρώτη έκδοση για την πρώτη έκθεση, συγγνώμη, ότι εδώ για 30 χρόνια αφήσαμε να αναπτύσσεται ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο στοχεύει μόνο στο κέρδος, χωρίς ηθική, χωρίς ηθικούς ενδιασμούς και οδηγεί σε, αυτούς, ε, σε αυτού του είδους τις ε, παρεκκλήσεις. Εγώ δεν θέλω όμως να δώσω αυτή τη μάχη μονάχη μου. Και δεν θα ξαναρχίσω την ίδια συζήτηση που έγινε στην, για την πρώτη έκθεση. Η βαθιά μου πεποίθηση για την ε, υπόσταση αυτής της κρίσης δεν έχει αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι τα δύο σημαντικότερα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν από την αρχή των εργασιών, της δεύτερης φάσης των εργασιών μας είναι δύο φαινόμενα που απορρέουν από την, από παρέκκληση του καπιταλισμού. Λοιπόν, εμείς θα συμφωνήσουμε άμα δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Για την προέλευση της κρίσης σίγουρα δεν συμφωνούμε, το είδα. Για τα offshore, για τους φορολογικούς παραδείσους, αν ας πούμε επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο παρεκκλήσεις, σίγουρα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Σίγουρα θα πρέπει να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης και για την Αραβική Άνοιξη, στην οποία έδωσα και σημαντική θέση ήδη, και για το τι γίνεται στη Ιαπωνία. Δεύτερη παρατήρηση που προέρχεται και από την ίδια δυσκολία που έχουμε στο να συνεργαζόμαστε είναι το θέμα της λιτότητας και της ηθικής. Αν δούμε τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, Ζητάμε μόνο από τους μισθωτούς να πληρώσουν τις επιπτώσεις μίας κρίσης που δημιουργήθηκε από τη συμπεριφορά των πρωταγωνιστών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μην μου λέτε ότι έγινε, το τι συνέβη στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία έγινε γιατί οι Έλληνες ή οι Πορτογάλοι είναι τεμπέληδες ή γιατί οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους. Και ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι δεν συμφωνείτε. Κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν συμφωνείτε, γι' αυτό την ξανανοίγω τη συζήτηση. Γιατί εγώ θέλω τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα μεταξύ μας. Ή θα, ή θα συμφωνήσουμε για να μην συμφωνούμε ή θα συμφωνήσουμε για να συμφωνήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό ο όρος για, τι για τις διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν θέλω ναι, αυτή η έκθεση να έρθει. Να έρθει παραμορφωμένη από τις τροπολογίες και οι Πορτογάλοι δεν θα καταλάβουν ποτέ τι θα λέει. Αλλά και οι τραπεζίτες δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και πέστε μας εσείς, τι κατάλαβαν οι τραπεζίτες λαδώνουν εδώ τους διάφορους συναδέλφους για να ψηφίζουν τελικά τα θύματα να είναι αυτά που πληρώνουν κάθε φορά που γίνεται κάτι. Εγώ ψάχνω να βρω ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να βγάλουμε τους Ευρωπαίους από την κρίση. Μα δεν μπορούμε να λέμε κάθε φορά ο λαός δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει, τι πρέπει να αλλάξουμε. Μα φυσικά δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά. Σίγουρα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να, να, ζούμε μόνο με ιδιωτικέ πιστώσεις, δεν μπορούμε να ζούμε με τα πυρηνικά, πρέπει να αλλάξουμε τρόπους κατανάλωσης, ότι οι, οι πόροι δεν είναι... Λοιπόν, ένα λεπτό. Διακόπτω, λέει συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν με κατάλαβε. Όταν είπα ότι δεν έχουν αλλάξει συμπεριφορέ, εγώ εννοούσα συμπεριφορέ των τραπεζιτών και τίποτα άλλο μόνο. Μα όταν μίλησε για τη συμπεριφορά των ε, διαφόρων πρωταγωνιστών και εγώ φαντάστηκα ότι μιλούσε για του τραπεζίτε. Αλλά επειδή στον απολογισμό ε, της αποστολής μας στην Αθήνα είπες ότι οι άνθρωποι δεν άλλαζαν. Μα όχι, εγώ πήρα το παράδειγμα της ε, Σουηδίας, όταν η Σουηδία αντιμετώπισε μια, αντιμετώπισε μια αντίστοιχη Κρήτη, α, και Φιλανδή και τότε είπανε Πρέπει να αφήσουμε παράμερα τις πολιτικές μας διαφορές, τις ιδεολογικές μας διαφορές. Είπανε λοιπόν η πολιτική είναι εθνική η κρίση. Πρέπει να τα βάλουμε λοιπόν όλα στο τραπέζι από κοινού. Και αυτό δεν συμβαίνει ούτε στην Πορτογαλία ούτε στην Ελλάδα. Το, αυτό δεν υπάρχει ούτε στην Πορτογαλία ούτε στην Ελλάδα λέει η κυρία Περέζη. Μα αυτό δεν είναι το αντικείμενο της έκθεσης γιατί αλλιώς δεν τελειώνουμε ποτέ. Αλλά τι προτείνουμε όμως στην Φιλανδία. Τι κάναμε στη Φιλανδία και στη Σουηδία και τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Εγώ πήγα στη ΔΟΕ την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη και ξεπλάγιν από δύο πολύ ε, σημαντικά επιχειρήματα του κυρίου Σωμαδία, του αφεντικού της ΔΟΕ, είπε για, το, για την αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας και το κόστος, το τομικό κόστος της εργασίας και με αυτό που μας είχε πει και ο Ζακ Τελόγο στη στο δείπνο με τους εθνικούς βουλευτές. Τι είπε. Όταν η Κομισιόν αναφέρει την αναπροσαρμογή των μισθών, την, την άτα των μισθών, Μα γιατί είχε εφαρμοστεί. Ήταν ένα στοιχείο προσαρμογής ε, των μισθών προς τους εργαζόμενους εκείνους που είχαν πληθωριστικές τάσεις, μισθολογικές πληθωριστικές τάσεις. Ο μηχανισμός λοιπόν της ΆΤΑ υπάρχει και έχει τις ίδιες αρετές. Και για την ανταγωνιστικότητα οι οικονομολόγοι της ε, ΔΟΕ λένε η ανάλυση της ανταγωνιστικότητας δεν, μάλλον η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντιφατική με την, τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Και όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή στην Ελλάδα, το πρόβλημα δεν είναι στην αξιολόγηση του μισθού, είναι στην αλυσίδα παραγωγής. Όταν εμείς παίρνουμε το ατομικό κόστος εργασίας ως πρώτο επιχείρημα για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, παίρνουμε το θέμα από την κακή του πλευρά. Και αυτό συνεχίζεται. Σήμερα τα έσοδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χρησιμοποιήθηκαν στην Ασία ή στη Λατινική Αμερική είναι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούνται είναι τριμερές όργανο η ΔΟΕ. Πάντως κανένας δεν έχει τη διάθεση να βιώσει την εμπειρία που βιώσαμε με την πρώτη έκθεση, αλλά ξέρω πολύ καλά που πατάω. Και τελευταία γενική παρατήρηση. Για τον φεντεραλισμό. Ήταν πολύ επίκαιρο το θέμα και ως Ευρωπαίοι έχουμε πραγματική ευθύνη. Όταν οι Ευρωπαίοι μιλάνε για την κοινοτική μέθοδο αναφέρονται στον κοινωνικό διάλογο, στο διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων στην κοινοτική μέθοδο και πρέπει αυτό να το θυμίζουμε. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε για τον δημοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας θα ήθελα να έχω τροπολογίες. Διότι εγώ τρομοκρατούμε όταν βλέπω τι συμβαίνει στη χώρα μου, τι συνέβη την Κυριακή. Το να μιλάει κανείς για Ευρώπη στις χώρες μας γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολο. Τι βλέπει ο κόσμος. Ότι η κρίση είναι εδώ και, έχει ριζώσει εδώ και τρία χρόνια. Και η Ευρώπη συνεισέφερε με αυτό που είχε να συνεισφέρει, με τη λιτότητα. Και να απαντήσω στον συνάδελφο Χουντή. Αυτό που προτείνω είναι το αντίθετο από την απλούστευμένη διαδικασία. Εγώ θέλω μία σύμβαση για να μιλάμε σαφώς για τα πράγματα και να προχωρούμε δηλαδή μέσα από μία ευρωπαϊκή κλίμακα που θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Και θα σταθώ τώρα σε άλλες απαντήσεις. Ο Έγγελς έφυγε, δεν χρειάζεται να το απαντήσω. Ανέφερε ένα σημείο όμως πολύ ουσιαστικό. Το θέμα των εργασιών των δημοσιονομικών της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικών Προοπτικών. Πρέπει να έχουμε και εμείς ορισμένες φιλοδοξίες για να μην διαχυθούν στις, άλλες, ε, στις εργασίες των άλλων επιτροπών. Φυσικά όμως στο πλαίσιο της εντολής μας. Ο Κοφεράτη έκανε παρατηρήσεις Είναι πολύ σημαντική η ιδέα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε επιλογές. Είναι ουσιαστικότατη, αλλά εμείς δημιουργούμε εδώ περιθώρια χειρισμών ζητώντας απλά και μόνο λιτότητα. Ή θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται για να χρηματοδοτήσουμε τις μελλοντικές επενδύσεις. Και αυτό φυσικά όχι μόνο με κινέζικα κεφάλαια που να χρηματοδοτούν δηλαδή μια ειφόρο ανάπτυξη για τους Ευρωπαίους. Ο συνάδελφος Σμιτ είπε και το σημείωσα και είπε ότι είναι απαγοητευτικό αν οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν. δεν... Αν, αν μιλούσε μόνο για τους Έλληνες, εγώ δεν συμφωνώ. Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν ορισμένα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι μόνο οι πιο φτωχοί που σφίγγουν το ζωνάρι. Όλοι πρέπει να αποφασίσουν ότι θα ζήσουν με λιγότερη κατανάλωση, με λιγότερη ενέργεια. Τώρα, το μήνυμα που αισθάνθηκα να βγαίνει από αυτή την Επιτροπή από την αρχή και δεν Κατάλαβα ότι οι νέες αλλαγές ε, στην κρίση άλλαξαν αυτή την προοπτική. Για τους G20 έχουμε και ένα συμβούλιο σχετικό στον... το οποίο συνεδρίασε και υπάρχει ένα πρόβλημα για την εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ. Αυτές όμως τις δομές ad hoc θα πρέπει να τις δούμε παράλληλα με τον ΟΙΕ. Η ιδρυτική αρχή της νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης πρέπει να περνάει μέσα από διεθνείς οργανισμούς και όχι μέσα από φόρουμ τα οποία δεν μπορούν να δίνουν συνέχεια σε αυτά που αποφασίζουν και είναι λίγο σαν σύριαλ που δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και δεν έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα και πρέπει να έχουμε όραμα. Αλλά πρέπει να λέμε ότι δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Το να εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το G20 δεν νομίζω ότι στέκει γιατί δεν, μπορεί να, δεν κρατάει τους λόγους του. Τώρα για τον Εγώ δεν θέλω να επανέλθω σε ζητήματα που αφορούν στην διάρκεια, στην ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα είχαμε συζητήσει στην πρώτη έκθεση. Ίσως βέβαια να υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να ξανανοίξουμε. Για το θέμα της παραγράφου 5 για τα έσοδα και την φορολογία. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αυτό μπαίνει λίγο και με τη, με τη συζήτηση για τον κύριο Ευρώ. Δεν τον έβαλα στην έκθεσή μου. Βλέπουμε τι γίνεται με την κυρία Άστον. Και το κείμενο πρεσβεύει την επιστροφή στην καθαρή κοινοτική μέθοδο. Η δυνατότητα πρωτοβουλίας, παρεμ, ε, ε, και επιβολής ε, ορισμένων επιτρόπων θα έπρεπε να αλλάξει. Εμένα η ιδέα μου που δεν έχει αλλάξει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρθρωση μεταξύ χρηματοπιστωτικών ε, αγορών και των αρμοδίων υπηρεσιών της, Ευρωπαϊκής, της Κομισιόν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από καιρό, δηλαδή ότι έναντι της κεντρικής τράπεζας δεν έχουμε κανέναν ο οποίος να αναλύει την κατάσταση ή να κάνει την αντιπραγματογνωμοσύνη. Αυτό που λέγει και ο Ντελόρ δηλαδή. Να προχωρήσουν τα πράγματα, να δοθούν νέα κίνητρα, μα αυτό κάνουμε όμως και εμείς σήμερα. Να υπάρχει μια ολοκλήρωση των οικονομικών πολιτικών και εγώ δεν ε, προσδοκώ να έρχεται όλη αυτή η εμπειρία η πραγματογνωμοσύνη μόνο από την Κεντρική Τράπεζα. Και υπάρχει το εξής παράδοξο, το πώς κοιτάζαμε εμείς πριν έρθει το ευρώ στις χώρες μας. Πώς τα βλέπαμε τα πράγματα για τις ισοτιμίες, για τη η υπερχρέωση του κράτους ή εθνικές κεντρικές τράπεζες το αντιμετώπιζαν το θέμα. Σήμερα όμως, αν πρόκειται για την Ελλάδα, την Πορτογαλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρώτα βασίζεται κανείς στην κεντρική τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα λοιπόν έχει μία εντολή που αφορά στην νομισματική πολιτική. Και αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε η Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που διευθύνει που θα, θα παίζει το δικό της ε, ε, θα, θα, θα, παίζει το, δικό της τροπάριο δηλαδή Αντί να ασχολείται τι γίνεται ας πούμε με τα ταμιευτήρια στη Γερμανία, με τις τράπεζες, με, το, με τη χρέωση ή δεν ξέρω τι, ασχολείται με το ύψος των μισθών. πλούστε την να θεώρηση της συνθήκης, εγώ ήμουνα κατά και έκανα και αποχή για τις τροπολογίες εκείνες που αφορούσαν στο θέμα και έπρεπε βέβαια να περάσουν αυτές ε, υπέρ των Ελλήνων και Πορτογάλων φίλων μας αλλά αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αναθεώρηση της συνθήκης χωρίς να υπάρχει ουστική δύναμη του Κοινοβουλίου για την αύξηση του χρέους και κοινωνικό ζήτημα. Αυτό το απάντησα προηγουμένως. Η Λίζα... Α, η κυρία Πίτικανεν λέει για την κοινοτική μέθοδο τι θέλει να πει αυτό και την κοινωτική τράπεζα. Ε, μα αυτό θέτει το θέμα της ε, δημοκρατικής ε, μεθόδου, είμαι ανοιχτή στις τροπολογίες, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό. Τώρα για την κρίση της δημοκρατίας της ε, κυρίας Γιάκων Σάρη. Όταν βλέπω τι γίνεται στην Πορτογαλία, μα πώς να πλήσετε κανείς που υπάρχει κρίση στην Πορτογαλία. Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο έχει απορροφήσει τέσσερα προγράμματα λιτότητας. Δηλαδή σε τρεις μήνες ένα πρόγραμμα λιτότητας έπρεπε να είναι επιτυχές για να μην το ακολουθήσει ένα άλλο. Μα αν δεν αφήσει κανείς τη χώρα ήσυχη για να μπορέσει να πάρει τα πάνω της αφού έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λιτότητας, πώς θα να σηκωθεί και για την κρίση της ε, δημοκρατίας. Ε, τι ζητάμε εμείς από την Πορτογαλία και τι τους δώσαμε από πριν. Πάντως σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ερμηνεύσατε ορθά τον όρο ακτέρ, τον όρο πρωταγωνιστής. Και χαίρομαι που σημερίζεστε κι εσείς ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές ακόμη δεν έχουν πάρει χαμπάρι για το τι σημαίνει κρίση. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη να απαντήσουμε για τον ευρωσκεπτικισμό. Σας απάντησα για τις ε, προτάσεις σας. Αυτοί που δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω αν θα το τραβούσα τόσο πολύ το σκηνή. Και εγώ είμαι πολύ ευρωπαίστρια όπως και εσείς. Αλλά η ευρωπαϊκή οικοδόμηση δεν στήθηκε έτσι. Και αν ας πούμε αύριο μας έρθει και η Τουρκία, θα πρέπει να φανταστούμε να συνεχίζουμε σε αυτήν την τόσο δημιουργική αμφισημία και αυτοί που είναι μέσα στη ζώνη ευρώ θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μακρηγόρησα, αλλά πραγματικά έπρεπε να πω ορισμένα πράγματα και μέσα από τις τροπολογίες δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να τα φύξουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ Περβάς και σένα και όλους τους άλλους συναδέλφους που συμμετείχαν. Δύο σύντομα σχόλια για το τέλος. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. 13η Απριλίου. Σας παρακαλώ μέχρι τότε να κάνετε τις τροπολογίες σας. Το αργότερο είναι Τετάρτη, 13 Απριλίου. Και επόμενη κοινή συνεδρίαση 11 Απριλίου στις 4 το απόγευμα θα έρθει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσης του Κογκρέσου από την Ουάσιγκτον να μας θα πει και στις 12 του μηνός έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε την περβάνς παραμονή της λήξης προθεσμίας των τροπολογιών. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπερές, ε, θα δεχόσασταν ε, να κατατεθούν οι τροπολογίες μόνο ε, υπό την αιγίδα των συντονιστών και των σκιωδών εισηγητών και όχι με μονομένες τροπολογίες. Ο καθένας στην ομάδα του να συντονίσει ε, με βάση τη μέθοδο που υιοθετήσαμε από την αρχή ε, του Δευτέρου Εμίσεως της θητείας. Ο Πρόεδρος. Θα το υποστήριζα αυτό προσωπικά, άλλωστε συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε τις τροπολογίες να τις κρατήσουμε περιορισμένες στον αριθμό και νομίζω ότι είναι και ρεαλιστική αυτή η πρόταση. Να κοιτάνε οι συντονιστές τις τροπολογίες της δικής τους πολιτικής ομάδας, να τις συνενώνουν και μετά ε, να τις υποβάλουν αφού τις έχουν χτενίσει. Εντάξει, λοιπόν, ε, ευχαριστώ. Ραντεβού στις 11 θα έρθει ο κύριος Αγγελίδης, πρόεδρος Επιτροπής Κρίσης του Κογκρέσου. Στις 12 του μηνός θα συζητήσουμε μαζί με την Περβάνς ε, και στις 13 λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ.